the floor. Good afternoon, everybody. Um, please can we adopt this afternoon's agenda? Αν θέλετε, εγκρίνουμε, λέει Πρόεδρος, την ημερησία διάταξη της σημερινής σας. και σας υπενθυμίζω ότι μεταδίδεται από το ίντερνετ η συνεδρίαση, οπότε παρακολουθούν και εκτός ε, συνεδριάσεως και υπάρχουν επίσης ε, στο ίντερνετ κάποια έγγραφα να δούμε τώρα κάποια άλλα θέματα πρακτικά. Έχουμε την ακρόαση σήμερα, δύο ενδιαφέρουσες ε, εκθέσεις, ψηφοφορίες και θα εξασφαλίσω την τήρηση των χρονικών ορίων, ούτως ώστε να τελειώσουμε στις 5. Άρα 5 παρατέταρτο το πρώτο κομμάτι και μετά ε, κάποιο διάλειμμα και μετά θα κάνουμε την ακρόαση, οι συντονιστές θα συνεδριάσουν αύριο στις 9.30. Κάνω και συνεδρίαση και κατόπιν θα κάνουμε την αξιολόγηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια επίσης με την Ήτρε, ε, Τζούρε και η Επιτροπή Γυναικών για την κυρία Γιώργα. Οπότε και αύριο υπάρχει πολλή δουλειά. Οπότε εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στα θέματα των συντονιστών ταχαίως αυτό πρόκειται να μας βοηθήσει πολύ. Και όλες οι συναντήσεις που σας είπα θα γίνουν σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Στο 6Q2. Can we approve the minutes from the previous meeting? Και να εγκρίνουμε τώρα τα πρακτικά από τις προηγουμένες συνεδριάσεις ή την προηγούμενη συνεδρίαση. Ωραία. Um, τώρα έχουμε τα το πρώτα πρώτα θέματα καταναλωτών, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πάρα πολύ επίκαιρο θέμα αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μέχρι τις 4 η ώρα και στη συνέχεια ε, το άλλο θέμα είναι οι ε, δυσμενείς διακρίσεις βάρος καταναλωτών στην ψηφιακή αγορά. Έχουμε τον κύριο Πατρισμούλιο από ε, το Λονδίνο, ο οποίο μα έχει ετοιμάσει αυτή τη μελέτη, θα προβεί μια παρουσίαση 10 λεπτών και αν κανεί ε, θέλει το λόγο, ε, σηκώστε το χέρι σα και θα σα γράψουμε στη σχετική λίστα ή κατάλογο. Θα σα πω τώρα με λίγα λόγια τι αφορά αυτή η μελέτη. Έχουμε και αυτέ τι διαφάνειε και οπότε να δούμε τώρα τα βασικά σημεία όπως θα φανιστούν στις διαφάνειες αυτές και τώρα όσο ετοιμάζεται η προβολή θα σας πω τι γίνεται. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε τι γίνεται όσον αφορά ε, τις υπηρεσίε υπηρεσίες και προστασία καταναλωτών ε, όταν ζητούν κάποιο προϊόν για να το ε, αποκτήσουν, να το αγοράσουν και στη συνέχεια δε να απαλληλωτριώσουν ούτως υπήν γενικώ το προϊόν για διάφορους τρόπους. Ε, έχουμε εδώ πέρα διάφορα προϊόντα στις υπηρεσίε υπηρεσίες και το βασικό θέμα είναι το ότι πολλές φορές όταν δεν έχουν σχετική εμπειρία δεν αγοράζουν κάποια προϊόντα οι καταναλωτές. Numerous market regulatory fails and there is potential for mis-selling. Να σας πω ότι εδώ τα θέματα δεν είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ σημαντικά. one of one of the uh, of the big ένα από τα θέματα που οδήγησαν στην κρίση ήταν τα στεγαστικά δάνεια, σχετικές ε, απάτες περί την ε, εκχώρηση αυτών των ε, δανείων. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύεται ο καταναλωτής και αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι να εξετάσουμε οι υπηρεσίες και αγαθά χρηματοοικονομικά που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους καταναλωτές ή για την νέα αγορά ή που να είναι ωφέλιμα για την ε, αγορά ή τους καταναλωτές μετά να δούμε κάποιο είδου ε, συμπεράσματα και κατόπιν συστάσεις. Όλα αυτά τα έχουμε βασίσει κάποιο είδου διαβούλευση με τους εμπλεκομένους και έτσι έχουμε του, τις ρυθμιστικές αρχές, ε, τους διαμεσολαβητές, τις ενός καταναλωτών, ε, τράπεζες, ε, ενώσεις τραπεζών κλπ. Να υποστιάσουμε προσοχή μας τώρα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα που ενδέχεται να είναι βλαπτικά. Τι εννοούμε βλαπτικά για καταναλωτές και μη έψιλον. Εννοούμε ότι αυτά τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, όταν κάτι πάει στραβά, τότε υπάρχει η πιθανότητα να βλάψουν την ε, τσέπη των καταναλωτών ή να τους ε, κάνουν πάρα πολύ βάλατους οικονομικά. οπότε θα να δούμε πότε σε ποιες πτώσεις υπάρχει παράτυπη πώληση ε, και τι γίνεται. Και για ποιο λόγο. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τους κινδύνους κατάλληλωτες ή καμιά φορά ε, υπάρχουν υποβολικά υψηλές δαπάνες, έξοδα, προμήθειες και με τέτοιου είδους ε, λεπτομέρειες ή με κάποια αντίστοιχα κίνητρα μπορεί κανείς να παγιδεύσει τον καταναλωτή τώρα δούμε ότι ποια προϊόντα συγκεκριμένα είναι αυτά. Πρώτα απ' είναι τα προϊόντα που έχουν σχέση με στεγαστικά δάνεια, ε, αυτά που είναι εκπεφρασμένα σε συνάλλαγμα ή μεταβλητού επιτοκίου και εδώ σας τονίζω και πάλι ότι δεν μιλούμε για πέντε ροδεκάρες Εάν ρίξετε μια ματιά στο τι είναι στην Ουγγαρία, εκεί υπήρχαν πάρα πολλά καταναλωτικά τα οποία ήταν υπερασμένα σε ευρώ και σε ελβετικό φράγκο. Και αν δείτε τι έγινε περί το 2007 και εάν υποθέσουμε ότι δεν είχαμε καμία υποτίμηση του Φιωρινιού, τότε ε, θα είχαμε 33%, θα έπρεπε να έχουμε 33% πιο μικρά, ε, πιο φτηνά στεγαστικά δάνεια. Είναι πολύ πιο ψηλά από το ΕΠ. Άρα βλέπετε ότι το άχθος που φέρνουν αυτού του είδους τα προϊόντα είναι πολύ σημαντικό. Επίσης έχουμε αυτές τις υψηλές προμήθειες, ιδίως όσον αφορά κάποια προϊόντα επενδυτικά, ε, σχετιζόμενα με συντάξεις και τέτοια. Έχουμε επομένως κάποια σύνταξη μετά από 46 χρόνια που είναι το βασική ηλικία, βασική διά, διάρκεια στην Αγγλία και οπότε πάνε για 5% που πληρώνουν σαν τόκο αντί για μισό της εκατό και τελικά θα έχουν απόδοση 33% λιγότερο. Επομένω 1% είναι η διαφορά στι ε, προμήθειε σημαίνει ότι έχουμε 33% λιγότερο ή μεγαλύτερο αντίστοιχα κόστος στο τέλος. Άρα βλέπετε ε, ότι μπορεί να φαίνεται ότι είναι μικρή διαφορά καταρχήν στην επιβάρυνση αλλά είναι πολλαπλάσιο η μεγαλυτερο αντιστοιχα κοστο στο τελο αρα βλεπετε οτι μπορει να φαινεται οτι ειναι μικρη διαφορα καταρχην στην επιβαρυνση αλλα ειναι πολλαπλασιο η επιβαρυνση των καταναλωτών. Τώρα δούμε πού προκύπτουν ζημιές για την ενιαία αγορά τι γίνεται τώρα με τους καταναλωτές, με τους όλους εμπλεκόμενους για συγκεκριμένα προϊόντα που μπορεί να την βλάψουν την αγορά, την ενιαία αγορά. Πρώτα-πρώτα ε, έχουμε πάρα πολύ ε, λίγες συναλλαγές οικονομικές διασυνοριακές και πρόσφατα μετρήσαμε ότι το 94% των καταναλωτών που δεν αγοράζουν στο εξωτερικό τέτοια προϊόντα θα το σκεφτόταν το 11% 94%. Επομένως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος δισταγμός να ψωνίσει κανείς στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν τα προϊόντα αυτά πολλούνται μόνο στο εσωτερικό της χώρας, τότε παρ' όλα αυτά μπορεί να έχουμε δυσμενείς στην ε, ενιαία αγορά. Ε, όταν οι επιπτώσεις είναι τόσο σημαντικές ώστε να εκείνο την ε, οικονομική σταθερότητα ή όταν έχουμε μια μεγάλη ομάδα καταναλωτών οι οποίοι επηρεάζονται και ε, αυτό επίσης έχει επιπτώσεις στα μη οικονομικά άγαθα και τις λοιπές αγορές επίσης υπάρχουν επιπτώσεις σε πολλούς καταναλωτές ακόμα και αν η κλίμακα για τον καθένα είναι μικρή. Οπότε αυτό ε, επιδρά και στην ροή του εμπορίου για άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες οπότε αυτά τα προϊόντα ε, αυτά τα συμβάντα γίνονται όταν έχουμε παράτυπη, παράνομη, αθέμητη πώληση όπως και τα ίδια όπως είπαμε και πριν τώρα να δούμε ποιες είναι οι υπηρεσίες και προϊόντα ε, είπαμε ότι είναι κάποια προϊόντα σε σχέση με στεγαστικά δάνεια που έχουν μεγάλες επιπτώσεις για τα φυσικά πρόσωπα αλλά και γι' αυτό το λόγο έχουν επιπτώσεις και σε ολόκληρε τι οικονομίε και σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, το διασυνορικό εμπόριο και αυτό το διαπιστώσαμε και εις την, στη ΣΥΠΑ αλλά και σε Ιρλανδία και Ισπανία. Τώρα έχουμε την ασφάλεια για προστασία της αποπληρωμής, ένα άλλο προϊόν το οποίο και αυτό μπορεί να φέρει πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις είναι πάρα πολύ καυτό θέμα τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τελευταίοι υπολογισμοί λένε ότι πάνω κάτω 28,8 δις στερλίνες έχουν ε, αλλάξει χέρια παράτυπα. 1,4% του ΑΕΠ της χώρας δηλαδή. Και αυτό το ποσό είναι τόσο γιγαντιαίο ότι όταν ε, να δώσουν κάποια αντιστάθμιση γι' αυτό η αποζημίωση αυτό ε, την αγορά σαν αυτοκινήτου γιατί όλοι είχαν στα χέρια πολλά λεφτά ε, γιατί σωρεύτηκαν αυτές οι αξιώσεις με τον καιρό επομένως βλέπουμε ότι μηνιαία το ποσό ήταν μικρό αλλά σωρευτικά το ποσό αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό Βεβαίω και έχουμε υπηρεσίε και τέτοια προϊόντα τα οποία είναι εποφελία των καταναλωτών και της ενιαίας αγοράς. Εδώ έχουμε κάποια τέτοια προϊόντα τα οποία είναι φτιαγμένα για τις ανάγκες του καθενός απλά, οπότε χρειάζεται αυτό το φτιαγμένο δηλαδή επιμέτρο το ΣΥΠΗΝ ε, είναι απλό και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στους καταναλωτές τότε να υπάρχει κάποια ευελιξία για τη διαχείριση του θέματος οπότε αυτό ε, συρρυκνώνει και τα έξοδα ε, όπως ας πούμε αυτά τα λεγόμενα consolidation loans, κάποια δάνεια. Θα σε εξηγήσω τι είναι αυτά τα προϊόντα, πάντως ε, προστατεύουν κάποιους που θα πτωχεύσουν ή εν όλο ή εν μέρη. Υπάρχουν πολλές απόψεις βέβαια, αλλά γενικώ είναι κάτι αυτά τα προϊόντα και επίσης είναι άλλα προϊόντα τα οποία διευκολύνουν τις ισορικές αλλαγές το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ε, χρεωστικές κάρτες, τις κάρτες και έχουμε όμως και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία ωφελούν τους καταναλωτάς όπως εδώ αυτά αποφελούν και την ενιαία αγορά, αυτά τα προϊόντα και τα οποία διευκολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο, την κινητικότητα των εργαζομένων, οπότε εδώ ο, ο βασικός τοπικός λογαριασμός είναι σημαντικός παράγον και αυτό έχει καταγραφεί ότι ωφελεί την κινητικότητα ε, σε σχέση με τις ε, υπηρεσίες πληρωμής, τα σχετικά δίκτυα Και εδώ έχουμε το ΣΕΚΙ ε, και την σχετική οδηγία. Αυτή η οδηγία για την καταναλωτική πίστη είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τις συναλλαγές της διασυνοριακές. Ποια είναι τώρα τα βασικά σημεία που μπορούμε να εξαγάγουμε εάν ανατρέξουμε στις αιτίες της κρίσης. Μια σημαντική αιτία ήταν κάποιο είδου αθέμητε πωλήσει, παράτυπες πωλήσει ε, κάποιων προϊόντων στεγαστικών δανείων. Και οι διαβουλεύσει έδειξαν ότι τα στεγαστικά δάνεια αφορούν τόσο μεγάλα ποσά που ήταν το πιο σημαντικό και για τα φυσικά πρόσωπα και για την γενικότερη οικονομική σταθερότητα. Μην ξεχνούμε επίσης ότι κάποια από αυτά τα προϊόντα τα οποία είπαμε ότι είναι βλαπτικά από την άλλη μεριά μπορούν να είναι και υποφελή. Άρα έχουμε δύο όψεις του ίδιου προϊόντος, του ίδιου νομίσματος άρα δεν είναι κάτι κακό αυτό. Επίσης βλέπουμε ότι τα θέματα αυτά έχουν ανακύψει και στη ΣΥΠΑ και στα κρατημέλη αλλά έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα προβλήματα με πρωτοβουλίες και του G20. Άρα βλέπουμε ότι έχει μπει ένα όριο στο πόσο κανείς μπορεί να χειραγωγήσει τους καταναλωτές σε αυτό το επίπεδο. Επίσης ήταν κάποια δεκαετία όπου είχαμε καινοτομίες, είχαμε απελευθέρωση αυτών των προϊόντων, παρ' όλα αυτά όμως οι καταναλωτές δεν έχουν τα προσόντα να διαχειριστούν αυτή την αγορά αυτά τα προϊόντα. Δεν λέω όλοι, αλλά η πλειοψηφία. Άρα χρειάζεται κανείς να είναι ενημερωμένος όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά. Και καταλήγουμε τώρα στο ποιες είναι οι προτάσεις, οι συστάσεις μας, οι οποίες εδώ είναι ομαδοποιημένες ανάλογα με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων. Πρώτα-πρώτα σημαντικός στόχος κατά μας είναι να μην υπάρχει ασυμμετρία πληροφοριών μεταξύ των παρόχων των υπηρεσιών αυτών και των καταναλωτών, γιατί ε, οι καταναλωτέ δεν αγοράζουν και τόσο συχνά, άρα έχουν πολύ λιγότερε πληροφορίε από αυτόν ο οποίο πολύ πλασάρει τέλο πάντων αυτά τα προϊόντα συνεχώ. Άρα πρώτα πρώτα θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίε συγκρίσιμε και ακριβεί. Άρα η οδηγία σε είναι πολύ σημαντική αλλά δεν αρκεί καλύπτει πάρα πολλές ε, πτυχές που έχουμε δει σε άλλες μελέτες όπου ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει καν τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου και του APRC. Άλλο. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το συναντούμε αυτό και σε άλλους τομείς, είναι να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες για τον μέσο καταναλωτή. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, Αυτέ οι ρυθμίσει για λέω ότι Να βρεθούν κάποια κριτήρια κατανοητά. Να, να, του πούμε ποιο είναι κάθε φορά το καλύτερο και το χειρότερο ε, σενάριο ακριβώς σαν τα επιτόκια των, ε, των στεγαστικών δανείων όπως κάποια δάνεια κοινωτικών αρχών όταν έχουμε κάποιο είδου υποτιμήσεις και πάντοτε να δίνονται παραδείγματα επεξηγηματικά. Πολλές φορές θα πρέπει να έχουν κάποιον ανεξάρτητο σύμβουλο καταναλωτές, να έχουν δυνατότητα να προσφύγουν, που να μην πολύ τίποτα ε, όταν μιλούμε για κάποια πολύπλοκα προϊόντα, γιατί οι καταναλωτές αυτά ε, δεν τα αγοράζουν συχνά, δεν ξέρουν. Άρα εδώ η συμβουλή είναι πάρα πολύ ε, σημαντική, Άρα πρέπει κάποιο χωρί να έχει εξαρτήσει ή σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, άλλες συστάσεις είναι οι εξής. πώς θα καταστούν τον καταναλωτή πιο ικανό να χειρίζεται αυτά τα θέματα. Είπαμε, γίνονται πολλές προσπάθειες, θα πρέπει να γίνουν περισσότερες και υπάρχουν και διάφορα προγράμματα, αλλά δεν υπάρχει αρκετή ζήμωση, δεν, δεν μια χώρα από την εμπειρία της άλλης ούτω ώστε να ξέρουν οι χώρε τι αποδίδει και δεν αποδίδει από αυτά τα μέτρα αυτέ τι πρωτοβουλίε. Επίση, του δίνουν πληροφορίε του καταναλωτή, τον εκπαιδεύουμε. Όμω παραμένουν και άλλα ζητήματα στην χρηματοοικονομική αγορά. Θα πρέπει ομένω να αναβαθμίσουν την προστασία του καταναλωτή. Από τι εξή απόψει. Πρώτα-πρώτα, εκ των προτέρων. Οι ρυθμιστικέ αρχέ θα πρέπει να είναι πιο ενεργές όσον αφορά να ερευνούν την αγορά. Εκ των προτέρων να ψάχνουν πού μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Πολλές φορές εκ των υστέρων μόνο παρεμβαίνει η ρυθμιστική αγορά. Άπαξ και προκύψουν τα προβλήματα. Τότε αναλαμβάνουν δράση οι ρυθμιστικές αρχές. Άρα για να μην υπάρχουν προβλήματα είναι σημαντικό να είμαστε πιο ενεργοί, πιο αποφασιστικοί να προστατεύουμε την αγορά και τον καταναλωτή από πριν. Οπότε αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και στην επαγόρευση κάποιων προϊόντων. Εάν θεωρεί η, η αρχή ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει κάτι ύποπτο και στο MIFID και στο MIFID 2 έχουμε ε, τέτοιες ε, ρυθμίσεις, τέτοιες προβλέψεις. Θα πρέπει βέβαια κάθε φορά να υπολογίζει ρυθμιστική αρχή το τι πρέπει να γίνει. Άλλα ζηματικά θέματα είναι ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να δουν εάν όλα είναι καλά με τις χρεώσεις, με τις ε, ε, προμήθειες, να μην είναι υπερβαλλόντως υψηλές αυτές οι χρεώσεις, ιδίως όσον αφορά κάποια μακροπρόθεσμα δάνεια, γιατί είπαμε ότι αυτό μπορεί να είναι σοπεδωτικό για τις συντάξεις, αν τα σχετικά έξοδα είναι τόσο ψηλά. Αλλά αυτό αφορά οποιοδήποτε μακρόπνο προϊόν. Τέλος, οι κυρώσεις. Οι κυρώσεις επιβάλλονται βέβαια εκ των υστέρων και αυτό θα πρέπει βέβαια να έχει και αποτελεπτικό αποτέλεσμα, όμως κανείς θα πρέπει να έχει ως σκοπό όχι μόνο να καταστήσει υπεύθυνο το χρηματοοικονομικό ίδρυμα το εκάστοτε, αλλά θα πρέπει αυτό να αφορά και κάποιους ε, υπαλλήλους όποτε έχουμε περιπτώσεις απάντησε. Και στην οδηγία αυτό προβλέπεται, αλλά θα πρέπει να ισχύσει και για τις λιανικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Επίσης, σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να προβλέπεται αποζημίωση του καταναλωτή. Βέβαια είναι με... μεγάλη συζήτηση για το πώς θα γίνει αυτό, ποιος θα είναι ο υπόλογος, υπεύθυνο γι' αυτό. Τώρα, τι γίνεται όποτε προκύψει το πρόβλημα, σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική ανεξάρτητη αρχή που έχει μηχανισμό επίλυση συναλλαγών που δεν κοστίζει πολλά ε, στις περισσότερες χώρες. Δεν υπάρχει διαμεσολαβητής για τα χρηματοοικονομικά. Επομένως, όταν έχετε μια τέτοια διαφορά με αυτόν που σας πωλεί κάποιο ε, προϊόν, ε, όταν πρόκειται για μεγάλο ποσό, μπορεί να μην θέλετε, να μην μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια. Άρα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να έχετε πρόσβαση ε, σε ένα εξοδικαστικό πλαίσιο και σύστημα. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει κάτι που να καλύπτει την ε, χρεοκοπία, την πτώχευση. Την υπερχρέωση ας πούμε και αυτό Γιατί δεν προβλέπει κάποιο μηχανισμό, αλλά θα έπρεπε να προβλέπεται και έτσι, να μπορεί ο, να σταθεί στα πόδια του ξανά ο καταναλωτή. Αλλιώ είδατε τι έγινε στην Ισπανία που κανεί δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του στεγαστικού δανείου εκτό εάν κατά κάποιο τρόπο ε, ως διαμαγείας η τράπεζα κάνει κάτι. Οπότε κανεί χάνει ποταμιεύσει που έχει επενδύσει, χάνει το σπίτι του και δεν μπορούν οι καταναλωτές ξανά να απολάβουν κάποιες χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Εδώ ολοκληρώσα την εισηγήσή μου και ευχαριστώ να σας απαντήσω τις ερωτήσεις Thank you very much, Mrs. Chairwoman. Ευχαριστώ. Μία από τις πρώτες συστάσεις που κάνατε ήταν η ενημέρωση για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, να είναι απλή και κατανοητή. Θα ρωτήσω λοιπόν, χρειαζόμαστε νέα νομοθετήματα για να επιτύχουμε αυτό το στόχο ή θα έπρεπε να το αναλάβει κάποιο, κάποιος ανεξάρτητος οργανισμός, πρόεδρος. Ε, νομίζω θα ακούσουμε δύο-τρεις ερωτήσεις και θα τα δούμε όλα μαζί καλύτερα. Κυρία ε, θα ήθελα σε σχέση με την έκθεση να μας πείτε ως προς την εμπειρία που είχατε στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, για τα μακροπρόθεσμα υψηλά επιτόκια και τις επιπτώσεις που είχε αυτό στην κοινωνία των πολιτών έχετε κάποια άλλα διδάγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο του χρόνου θα θεσπιστεί νέα νομοθεσία κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξοι μπορείτε να σχολιάσετε τα όρια για τα βραχυπρόθεσμα εξαιρετικά ε, υψηλά επιτόκια παραδείγματος χάρη η κυρία Στήλε, ε, για τα τέλη και για τις επιπρόσθετες επιβαρύνσεις ε, μας μιλήσατε στην έκθεσή σας. Ήθελα να πω ότι σημειώνονται πολλές εξελίξεις στην αγορά. Θα μπορούσατε ίσως να σχολιάσετε ε, τις βασικές, ε, κατά τη γνώμη σας, αλλαγές που έχουν γίνει, ώστε να μπορέσουν ε, απλούστερα, γρηγορότερα να αποπληρώνουν τα χρέη τους οι καταναλωτές, μήπως υπάρχουν, υπάρχουν και συγκεκριμένε απόψεις για αυτές τις ιστοσελίδες όπου γίνεται σύγκριση των διαφόρων δανείων, εξαρτάται βέβαια και από τις ανάγκες των καταναλωτών και αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ε, στην σελίδα 50, τώρα το σχολιάσατε αυτό το ζήτημα, ε, αυτό της διαφήμισης, ε, υπάρχει και ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός που μιλάει για τη διαφήμιση στα παιδιά για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. για τις ασφάλειες θα ήθελα να μας πείτε τι πιστεύετε για τις προτάσεις για τη διαμεσολάβηση στον τομέα των ασφαλιών ε, και τέλος ε, ε, για τον Λόρδο Χίλ τι σχόλιο θα είχατε να κάνετε σε σχέση με τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές δηλαδή τι θα προτείνατε εσείς στην επόμενη πενταετία να κάνει ο Λόρδος Χίλ σε αυτό το τομέα Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις και μετά θα κάνουμε και ένα άλλο δεύτερο γύρο εκτός μικροφώνου. Ε, νομίζω ότι είναι διαφορετική η κατάσταση από χώρα σε χώρα σε σχέση με την ε, κατανόηση αυτών των ζητημάτων. Οπότε ε, πολύ αυστηρή νομοθεσία και λεπτομερής νομοθεσία, δηλαδή ότι πρέπει να εξηγείται και να ενημερώνεται για το τάδε και για το δίνα, δεν νομίζω ότι ενδείκνεται. Ε, θα πρέπει ο πάροχος και ο νομοθέτης να έχουν ξεκαθαρίσει τι συνιστά ε, κατανοητή ενημέρωση. Δηλαδή, άμα έχετε 20 σελίδες πυκνογραμμένες, κανείς δεν πρόκειται να ενημερώσει αλλά παρόλα αυτά θα έχει υπογραφεί το, δάνειο και θα είναι αργά. Θα πρέπει για την συμπεριφορά να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, λεπτομερείς. Αυτά περιμένουμε από τον πάροχο, αλλά όχι για την εφαρμογή τώρα. Μπορούμε να δούμε ε, πώς αντιδρούν και οι καταναλωτές οι ίδιοι για τις διάφορες προτάσεις για την ετικετοθεσία. Παραδείγματος χάρη το έχουμε κάνει, γιατί όχι και εδώ. Ε, για τα, τα, τις ε, πιστώσεις ε, υψηλού κόστους που χορηγούνται άμεσα, δεν αναφέρθηκα σε αυτό, όντως υπάρχει μια σχετική αναφορά μέσα στην έκθεση, υπήρχε σοβαρή έλλειψη κατανόησης, δεν καταλάβουν οι γιατί πράγμα δεσμεύονταν Ορισμένε φορές πλήρωνε κάποιος 4.000 σαν τόκο και είναι πολύ σύντομο το δάνειο, κρατά τρεις ε, μήνες 4.000 ε, στις 100 μάλλον, όχι 4.000 πλέον, 4.000 στις 100 ήταν η επιβάρυνση, αφήστε τους τόκους υπερημέρειας. Ε, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπατε, αναλαμβάνει πολλά μέτρα για να περιορίσει τις δραστηριότητες αυτού του χρηματοπιστωτικού τομέου και σε σχέση με τις τελευταίες εκτιμήσεις, σε τρεις πάροχοι μόνο θα επιβιώσουν με την εφαρμογή ε, των νέων κανόνων, ε, μεταξύ των οποίων είναι και το όριο για το ανώτατο όριο για τα επιτόκια. Τι γίνεται κάποιο κάποιος χρειάζεται βραχυπρόθεσμα ένα δάνειο δύο-τρει μήνες ε, επειδή δεν υπάρχουν ε, πάροχοι που να δίνουν τέτοια προϊόντα. Δεν πρόκειται καμία τράπεζα να σα δώσει δάνειο για κάτω από 12 μήνες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια κατάσταση θα δημιουργηθεί στην αγορά και αν θα επιστρέψουν έτσι οι καρχαρίες και το κογλίφι στην αγορά ανάλογα με την, τα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί. Δηλαδή, άμα υπάρχει ζήτηση και θα υπάρχει ζήτηση για βαρχιπρόθεσμα δάνεια ε, έως τρεις μήνες, ε, ε αναμένεται να δούμε ποιο, πώς θα καλυφθεί αυτή η ζήτηση. Αυτά. Όχι. Για την ε, αυξημένη, αυξημένη διαφάνεια για την ενυπόθηκα. Ε, νομίζω ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η κατανόηση από πλευρά των καταναλωτών των πληροφοριών που ε, προσφέρουν οι πάροχοι. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δοκιμάζουν, να συμμετρούν την κατάσταση εξ άντε οι νομοθέτες ως προς τους νέους κανόνες για την ενημέρωση. Δηλαδή, ε, να, ε, ε, undercover να πηγαίνουν, να προσποιούνται ότι είναι καταναλωτές και να δοκιμάζουν τα προϊόντα. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε αν είναι αποτελεσματική η εφαρμογή. Θα περάσουμε από την εφαρμογή στην αποτελεσματική εφαρμογή. Μιλήσατε για τις που συγκρίνουν τα δάνεια. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, διότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο το ζήτημα, εάν δηλαδή δίνουν όντως συμβουλές ή όχι, εάν ε, είναι, ισχύουν οι πληροφορίες ή όχι, Για αυτές τις ε, ε, ιστοσελίδες ε, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως συνδέεται με ένα πάροχο. Αυτό μας υποδεικνύουν οι νομοθέτες και δεν το αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής διότι φέρει άλλη επωνυμία η εταιρεία, άλλη για την εταιρεία που δίνει τα δάνεια, άλλη για την ιστοσελίδα σύγκρισης. Οπότε δεν είναι, ε, ανεξάρ... Ε, δεν είναι αντικειμενικές οι πληροφορίες, αλλά απλώς αυτό εκφεύγει λίγο του πεδίου εφαρμογής της πρότασης. Γι' αυτό δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Ως προς την πρόοδο που σημειώθηκε, δεν είναι ξεκάθαρο ε, για τα επενδυτικά προϊόντα για τις ασφάλειες ζωής. Α πάρουμε αυτό είναι πολύ περίπλοκο το προϊόν. Δεν πρόκειται για προϊόντα, δηλαδή η ασφάλεια για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι. Ε, συνδέεται με ένα ε, συγκεκριμένο προϊόν η πρώτη κατηγορία και είναι πιο κατανοητό για τους καταναλωτές. Όταν περνάμε τώρα σε, ασφάλεια, σε επενδυτικά προϊόντα για την ασφάλεια ζωής, διότι είναι μεγάλη περίοδο ορίμανση, η περίοδος ορίμανσης μέχρι να αποβιώσει κάποιο Παραδείγματο παραδείγματος χάρη, ε, υποτιμάται το, ο κίνδυνος ε, που αναλαμβάνει κάποιος όταν προσυπογράφει ε, ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ο νομοθέτης σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο δηλαδή να μεριμνήσει ούτως ώστε οι πάροχοι να συμμορφώνονται με το πνεύμα των διατάξεων σχετικής οδηγίας για την βασική σύσταση που θα απίφθηνα στο Λόρδο Χίλ θα έλεγα όλα τα προηγούμενα δηλαδή ε, στην εξάντε εφαρμογή θα χορηγούσα περισσότερα κονδυλία δηλαδή να βγει στην αγορά ο νομοθέτης και να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή να μην περιμένει να προκύψουν τα προβλήματα διότι όταν ανακύπτουν τα προβλήματα πολύ συχνά έχουν πληγεί ή επιμολυνθεί α το πω έτσι πολλοί καταναλωτές ε, οι εξάντε προσέγγιση, εκ των προτέρων προσέγγιση είναι αυτή που θα προέκρινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι όντω αυτή η μελέτη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και βεβαίω, αναλύοντας την κάθε χώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλέ αρνητικές επιπτώσει. πολλοί καταναλωτέ πλήττονται από αυτέ τι ανισορροπίες που υπάρχουν και τι αναφέρατε βεβαίω και εσεί. Υπάρχει λοιπόν ανισορροπία μεταξύ των πληροφοριών που έχουν οι πληροφορίες, που έχουν ε, καταναλωτές και των ε, πληροφοριών που δίνουν οι υπάροχοι. Δεν κατάλαβα όμω κάτι από την έκθεση αυτή και ίσω θα μπορούσατε εσεί να μου πείτε κάτι. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να επιτύχουμε το εξή. Οι καταναλωτέ μα να καταλαβαίνουν καλύτερα τι πληροφορίε που λαμβάνουν. Ίσως θα πρέπει ε, κάπω πιο διαρθρωμένα να προχωρήσουμε εκ μέρου των ε, χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Ε, ε, ίσως να πρέπει να υπάρξει κάποιο, κάποιο βήμα, κάποιο σύστημα μέσα στο οποίο θα μπορεί να μπει ένα καταναλωτή και να ενημερωθεί, να λάβει τι πληροφορίε που χρειάζεται. Και από την άλλη, υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα που έχει κανείς να ε, διαπραγματευτεί. Ο παρόχος φυσικά έχει μεγαλύτερο πεδίο ευελιξίας ε, από αυτόν που πιέζεται και χρειάζεται εκείνη τη στιγμή τα χρήματα. Και από την πρακτική βλέπω και γνωρίζω πάρα πολλές περιπτώσεις όπου ανεξάρτητη σύμβουλοι μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Ξέρω πολλά παραδείγματα δηλαδή όπου αυτη η ανεξαρτητη τριτη άνθρωποι τελικά αυτό που κάνουν δεν βοηθάει τους καταναλωτές παρόλο που ο αρχικός τους ρόλος είναι αυτός αλλά αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά να το αποσπούν ακόμη περισσότερα χρήματα πιέζοντάς τον. Ίσως λοιπόν και εκεί από θεσμική άποψη θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει ανεξάρτητες πληροφορίες, αντικειμενικές πληροφορίες για να μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους τραγωδίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τη συνάδελφο και εγώ θέλω να μιλήσω για αυτά τα προβλήματα που ανέφερε η κυρία Γκραπίνη μόλις. Τι κάνουμε με την ε, εφαρμογή. Είπατε και εσείς ε, στην παραμβασή σας ε, ότι πολλοί πολίτες δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς γίνεται στα οικονομικά θέματα. Πολλοί, όπως είπατε, δεν γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει ακριβώς αυτό που γίνεται. Και τελικά κανείς δεν ξέρει στο τέλος αν ο καταναλωτής έχει λάβει όλες τις πληροφορίες και αν τις έχει καταλάβει ακόμη και να τις έχει λάβει. Ένα θέμα λοιπόν είναι να λάβει ο καταναλωτής πληροφορίες, ένα άλλο είναι να καταλάβει τις πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσει να τις αξιολογήσει. Αν τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα ε, με την εφαρμογή, ποιος έχει δίκιο τελικά. Αυτός που εξηγεί, γιατί αυτός θα πει, μα εγώ έδωσα τις πληροφορίες, άρα εγώ έχω το, είμαι, δίκιο με το μέρος μου αυτό το πρόβλημα πώς μπορούμε να το λύσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπου ίσως ε, εσείς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε, γιατί είπατε και εσείς ο ίδιος ότι μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Έχετε κάποια παραδείγματα να μας πείτε για το τι είναι αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Eh, Ευχαριστώ. Και εγώ θα συνεχίσω να θέτω ερωτήματα, όπως και οι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση της ε, μελέτης και για τις συστάσεις που μας κάνατε. Πραγματικά με εξέπληξαν οι συστάσεις που κάνατε σχετικά με την αύξηση της ε, ανεξαρτησίας ή της ε, πρόσβασης σε ανεξάρτητες πληροφορίες. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό, Πώς, πώς είναι δηλαδή μια ανεξάρτητη συμβουλή που δίνεται σε κάποιον. Και εκτός αυτού, όταν μιλούμε για, την, για το κατά πόσο καταλαβαίνουν ή όχι οι πολίτες τις πληροφορίες, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το να καταλαβαίνει κανείς ε, τα οικονομικά στοιχεία δεν επηρεάζει μόνο τις οικονομικές ή χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει ε, και οι πολίτες να καταλάβουν ε, ότι και οι πάροχοι έχουν τη δική τους ευθύνη βρίσκονται όλοι σε έναν φαύλο κύκλο γιατί πρέπει να πάρει κάποιος ένα δάνειο, να καλύψει ένα άλλο δάνειο που έχει πάρει και ουσιαστικά δεν καταλήγει πουθενά αυτή η ιστορία. Εσείς θεωρείτε ότι είναι δυνατόν οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε όσους ετούνται για να πάρουν ένα δάνειο να, να δίνονται με κάποιο πρότυπο τρόπο. Ευχαριστώ. Και να κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα γιατί δύο χρόνια τώρα ασχολήθηκα με την οδηγία για τα ανυπόθηκα δάνεια και είναι σημαντικό να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Τονίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά πρέπει να τονίζουμε και τα όσα έχουν γίνει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ψηφίσει λοιπόν ένα νομοθέτημα για, τις, ε, για τα ανυπόθηκα δάνεια, το οποίο εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη ας πούμε τα δάνεια ήταν υπόθηκα δάνεια τα οποία εκδίδονται σε άλλο νόμισμα, ε, οι πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες και βεβαίως η ανταλλαγή των πρακτικών από τα κράτη-μέλη, το θέμα των ενδιαμέσων επίσης είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε και τι έχουμε κάνει πριν αρχίσουμε να λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη νομοθεσία. Γιατί Επίσης υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες μα λένε ότι η πρόσβαση σε δανειοδότηση τώρα είναι πολύ δύσκολη. Ναι βεβαίω πρέπει να δράσουμε περισσότερο. Έχουμε κάνει όμως πάρα πολλά και με βάση τα μαθήματα που πήραμε από την κρίση. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε πρόσβαση σε δανειοδότηση. Εδώ μιλάμε για θέματα ενιαία αγορά. και κάποια από τα θέματα που αναφέρετε ίσω είναι θέματα εθνική αρμοδιότητας και αυτό είναι το πρόβλημα τη ισορροπία που πρέπει να έχουμε. Πότε ένα θέμα είναι ευρωπαϊκό και πότε είναι ε, εθνικό. Γιατί βεβαίω δεν θέλουμε να αρχίσουμε να αποσύρουμε τη δυνατότητα διατηνιοδότησης από κάποια μέρη, κομμάτια της αγοράς, υιοθετώντα τους ίδιους κανόνες, όταν θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει το θέμα αυτό αντιλάσσοντας απλώς βέλτιστες πρακτικές. Οπότε αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι αν όντω δουλεύουν, αν όντω ε, εφαρμόζεται καλά η ε, νομοθεσία γιατί είναι και καινούριο νομοθέτημα. Ε, υπήρξαν βεβαίω κάποιε ανησυχίε ότι κάποια από τα θέματα τυποποίηση των πληροφοριών θα μπορούσαν ίσω να επισύρουν μεγάλο κόστο για, για τον κλάδο. Έχουμε τελικά την, ισορροπία, την ε, αυτή που θέλαμε, να έχουμε τι σωστέ πληροφορίε χωρί να επιβαρύνουμε με περισσότερο κόστο. Και επίση, έχουν υπάρξει σκάνδαλα για καταχρήσεις, αλλά αυτό το θέμα είναι θέμα ενιαίας αγοράς. Μήπως είναι θέμα αποκλειστικά του κάθε κράτους μέλους. Δηλαδή υπάρχουν αποδείξεις ότι μιλάμε για τέτοιες καταχρήσεις διασυνοριακές, που πάνε από χώρα σε χώρα. Είναι όμως αυτό θέμα της ε, ενιαίας αγοράς. Και επίσης ε, οι όροι και οι προϋποθέσεις που υπάρχουν, ε, τα μικρά, τα ψηλά γράμματα, για, την, ε, για τα online όμως ε, ε, συμβόλαια που κάνουμε, αν κάποιος αγοράσει κάτι online ας πούμε, κάποιος σου ζητάνε απλώς να βάλεις ένα τικ σε ένα κουτάκι. Δεν διαβάζει κανένας τι, τι γίνεται πίσω από αυτό. Οπότε ίσως να πρέπει να δούμε και τα αγορέ και online αλλά και offline. Αυτό το που με ενδιαφέρει όμως εμένα είναι πότε μπορούμε να έχουμε δράσεις που από τη της και πότε μπορούμε να έχουμε και εθνικέ δράσεις που θα προστατεύσουν τον καταναλωτή αλλά θα του δώσουν ταυτόχρονα και πρόσβαση στη δανειοδότηση γιατί μα το λένε πάρα πολύ αυτό. Να ξεκινήσω απαντώντας στις τελευταίες σας ερωτήσεις. Έχουν γίνει όντω πολλά μέσω τη οδηγία για, για τα ανυπόθηκα δάνεια. Και αυτό είναι βεβαίως ε, σημαντικό. Το θέμα είναι πότε, πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Γιατί είναι σημαντικό ότι τα ε, δάνεια που εκδίδονται σε, σε άλλο νόμισμα είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά Αυτό, δεν, το πώς θα το λύσουμε δεν το ορίζει η ε, οδηγία. Είναι κάτι που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Και εγώ γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει και οι ρυθμιστές να βγούνε και να δούνε πώς εφαρμόζεται η οδηγία. Όλα αυτά που λέει η οδηγία, το πνεύμα της οδηγίας ε, υιοθετήθηκε. Γιατί ούτω ή άλλω το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Δεν μπορεί κανένα να εξηγήσει με απλά λόγια τον κίνδυνο. Είναι σημαντικό λοιπόν οι καταναλωτέ να έχουν μια σαφή εικόνα για το τι μπορεί να του συμβεί παίρνοντα ένα δάνειο. Α πούμε, παίρνει κάποιο ένα δάνειο εν υπόθηκο. Οποιοδήποτε μπορεί να πάρει ένα τέτοιο. Με την προπόθεση ότι αν δεν πληρώσει ε, τακτικά, δεν πληρώνει, μπορεί να χάσει το σπίτι σου. Όλοι λένε «Ε, εντάξει, εντάξει, δεν πρόκειται εμένα να μου συμβεί αυτό, εγώ θα πληρώνω. Ε, είναι ανθρώπινο αυτό. Αλλά όταν κανεί μιλήσει σε κάποιον, μπορεί ας πούμε, να του πει ότι μπορεί να είσαι άνεργο σε λίγα χρόνια, μπορεί να μην μπορεί να πληρώσει. Μόνο τότε αρχίζει κανεί να συνειδητοποιεί ότι δεν είναι κάτι σαφέ ή αφηρημένο το να μην μπορεί κάποιο να πληρώσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό το πώ το παρουσιάζουμε. Συμφωνώ ότι ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να υπάρξει μια γενική σύσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λέει ότι οι ρυθμιστέ θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια ε, προσέγγιση εξάντε, είναι λίγο πιο δραστήρια από την αρχή. Τώρα για το online και τα offline, ε, τις online και offline αγορές. Ε, ναι, είναι βεβαίως πολύ πιο ευρύ θέμα αυτό και δεν επηρεάζει μόνο τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ούτως ή άλλως ε, ε, μιλάμε για παντός είδους προϊόντα και υπηρεσίες και σίγουρα οι πολίτες, οι περισσότεροι δεν, δεν ξέρουν, έχουν ιδέα για το τι όρους και, και προϋποθέσεις έχουν εν αγνία τους δεχτεί. Τώρα για την ε, για τις ε, συμβουλές ε, για την κατανόηση, την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών αυτών στοιχείων. Για τα περίπλοκα προϊόντα, ας πούμε, τις υποθήκες με κειμενόμενο επιτόκιο, αυτά θα μπορούσαν ίσως να εμπέσουν σε μια τέτοια διαδικασία ή για κάποια επενδυτικά προϊόντα. Κυρίως όταν έχουμε θέματα όπως τα swaps. θα ήταν μάλλον πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή να έχει κάποια οικονομική συμβουλή αυτό το θέμα, πώς ε, μπορεί κανείς να το πληρώσει. Δηλαδή δεν μπορεί κανένα να υποχρεώσει τους παρόχους. Οι παρόχοι είναι ε, υπεύθυνοι να παρέχουν σωστές και αντιληπτές ε, συμβουλές στον καταναλωτή. Αυτό είναι μία προσέγγιση. Αν αυτό αρκεί, δεν ξέρω. Εμένα, εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες, γιατί πάντα υπάρχει και το θέμα του πώς εξηγεί κάποιος όλα αυτά σε έναν καταναλωτή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε και βεβαίως αυτό ίσως να αγγείται στην δικαιοδοσία των κρατών μελών περισσότερο αντί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει ένα σύστημα παροχής συμβουλών, συστάσεων, το οποίο θα μπορούσε ε, όπως, να είναι όπως το Ηνωμένο Βασιλείο, ε, το, που πληρώνεται από κάποια τέλη για τις, ε, για τις συμβουλές που παρέχει. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε τη δημιουργία ενός τέτοιου μοντέλου ή ένα μοντέλο για συμβουλές για, τη, για χρέος. υπάρχει αυτό, το fair share ας πούμε στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο από κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από τους παρόχους ηλεκτρισμού ή αερίου δίνουν ένα ποσό από τα έσοδά τους σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι συμβουλές, αυτή η παροχή συμβουλών ε, σε καταναλωτές χωρίς αυτοί να χρειαστεί να πάρουν έναν ιδιωτικό ε, πάροχο τέτοιων ε, συμβουλών. Οπότε ίσως καλό θα ήταν και κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει από μόνο του πώς μπορεί να το εφαρμόσει αυτό. Αλλά το θέμα το γενικότερο που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι αν γίνεται κάτι, αν, αν κινείται κάτι, αν υπάρχουν δηλαδή τέτοια μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι ότι όντω είναι καλά πληροφορημένοι οι καταναλωτέ. Αν τώρα είναι μόνο οι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και οι πάροχοι που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό, που είναι και αυτό μια πιθανή λύση, τότε νομίζω ότι η σύστασή μου προς τον Λόρδο Χίλ είναι πολύ σημαντική να ξεκινήσει δηλαδή αυτές τις εξάντε, αυτούς τους εξάντε ελέγχους. Αυτά, Πρόεδρε. Thank you. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για την ίδια, για την εφαρμογή, έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. second um, study is Δεύτερη μελέτη, ε, διακριτική ε, ε, αντιμετώπιση των πολιτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Έχουμε εδώ τον ε, καθηγητή αστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Όσνοβρουκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Very much, um, also for pronunciation. Um, I'm afraid my... Ευχαριστώ. Ε, ωραία το προφέρατε. Όχι τόσο καλά όσο θα προφέρω, ή μάλλον πολύ καλύτερα από θα προσφέρω εγώ τα αγγλικά τώρα. Τέλος πάντων θα μου πείτε μετά. Ε, ε, κάναμε μία μελέτη για την προηγούμενη επιτροπή, ε, ε για την προηγούμενη δηλαδή κοινοβουλευτική θητεία, ε, για την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Ο καταναλωτή είναι τόσο θαραλέο ε, που σε μια διασυνοριακή κατάσταση, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, πάει να κάνει παραγγελία εκτό τη χώρα του, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και συνειδητοποιεί ότι δεν γίνεται να την κάνει την παραγγελία ή ότι ισχύουν άλλες ε, προϋποθέσεις, άλλοι όροι σε άλλες χώρες. Λοιπόν, ε, εξετάσαμε το τι γίνεται στην πράξη, στο πραγματικό κόσμο. Και εστιάσαμε την προσοχή μας στο κείμενο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση διακριτικής μεταχείρισης για τους καταναλωτές και κάναμε κάποιες προτάσεις για την προστασία των δεδομένων που σίγουρα εσείς γνωρίζετε. 75% των πολιτών Λιανικής δεν ε, πολλούν διασυνοριακά σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό ισχύει με κάπως χαμηλότερο ποσοστό για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τα ε, δύο τρίτα των επιγραμμικών καταστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ποτέ δεν πολλούν πέραν των συνόρων. 9% μόνο των καταναλωτών στην καλύτερη περίπτωση αγοράζει ε, επιγραμμικά από κάποιο άλλο κράτος μέλος περίπου 50% στις φορές 55 και 60, 50% των διασυνοριακών πωλήσεων δεν έχουν ε, ευτυχή κατάληξη ή να το πω ανάποδα 15% μόνο έχει κάποια ευτυχή κατάληξη. Ποια είδη διακριτικής μεταχείρισης υπάρχουν. Ναι. Ε, άρνηση καταγραφής της παραγγελίας λόγω της γεωγραφικής θέσης, του τόπου διαμονής αν θέλετε, των καταναλωτών. Λένε στον καταναλωτή δεν πολλούμε στη χώρα σας. Επίσης, περιαγωγή ε, Δηλαδή ο καταναλωτής μπαίνει στην ιστοσελίδα που τον ενδιαφέρει, αλλά επανακατευθύνεται αυτόματα σε ένα υποκατάστημα του ίδιου παρόχου που όμως είναι εγκατεστημένο στο δικό του ε, κράτος μέρος, εκεί όπου διαμένει. Ε, όπου τα προϊόντα, η ποικιλία δηλαδή προσφέρεται ε, είναι διαφορετική, είναι υψηλότερες οι τιμές όπως δυστυχώς ανακαλύπτουν οι καταναλωτές, ισχύουν άλλοι όροι για την τιμολόγηση, παραδείγματο χάρη, που είναι εξαιρετικά ενοχλητικό. Δηλαδή, εγώ ξαφνικά ανακαλύπτω, α, ε, για μένα είναι ακριβότερο από ότι για τους καταναλωτές που βρίσκονται αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται η αυτή η εκτροπή λοιπόν των καταναλωτών και κάτι άλλο πολύ ενοχλητικό Εάν θέλετε να αγοράσετε ψηφιακό περιεχόμενο, ανακαλύπτεται ότι υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί χρήσης. Δεν μπορεί κάτι να, ε, που έχετε αγοράσει να το δείτε στη Γαλλία, παραδείγματο χάρη. Και είναι επαχθή στη διαδικασία για να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σα σε κάποια άλλη χώρα. Όμω, αν επιστρέψετε στην πρώτη χώρα που έγινε η αγορά, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχετε τέτοιου είδους προβλήματα έχουμε στην ψηφιακή εσωτερική αγορά. Ποιοι είναι οι λόγοι. Ε, είναι πολύ και διάφοροι. Κάποιοι είναι, ε, ανακοινώνονται επίσημα, κάποιοι άλλοι όχι. Ε, δεν σχετίζονται όλοι ε, με την παράδοση των προϊόντων, εφόσον μιλάμε ω επιτοπλίστων για την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Όμω ε, υπάρχει θέμα με τις πληρωμές παραδείγματο χάρη, την εφαρμογή τη σχετική διαδικασία. Υπάρχουν γλωσσικά, γλωσσικοί φραγμοί, παραδείγματος χάρη, όταν υπάρχουν καταγγελίε, ζητούνται οδηγίες σε μια γλώσσα που δεν προσφέρει η εταιρεία, παραδείγματο χάρη ε, στον κατάλογο των ε, δημοσιοποιημένων λόγων ε, υψηλή θέση έχει η νομική ασφάλεια. Θα επανέλθω σε αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Συχνά λένε οι επιχειρήσεις υπάρχουν άλλες προτιμήσεις στους καταναλωτές σε άλλες χώρες και για λόγους marketing επιθυμούμε να έχουμε ένα τοπικό ε, κατάστημα για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους καταναλωτές. Ε, φυσικά δεν αποκαλύπτουν ότι ε, σε ορισμένες χώρες τιμολογούν ακριβότερα τα προϊόντα. Για να δούμε τώρα το τωρινό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν μας βοηθάει πολύ το τωρινό πλαίσιο. Και όχι μόνο δεν μας βοηθάει, είναι και χειρότερα τα πράγματα. Υπάρχουν εγγενείς περιορισμοί ως προς το θεμελιώδες δικαίωμα της επιχείρησης που συνιστά από μόνο του φραγμό για την εφαρμογή της ομοθεσίας και την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης που υφίστανται οι καταναλωτές. Λοιπόν, εγώ θα ε, μπω σε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για την οδηγία για τις υπηρεσίες και θα αφήσω το υπόλοιπο ζήτημα ε, ε Βρυξέλλες 1, Ρώμη 1, δίκαιο ανταγωνισμού, πνευματικά δικαιώματα, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Όλα αυτά τα ζητήματα τα αφήσω να, για να μου υποβάλλετε εσείς συγκεκριμένα ερωτήματα, αν συμφωνείτε. Για να δούμε τώρα. Ε, το πρώτο που μας έρχεται ε, κατά νου είναι τα ατομικά δικαιώματα για την ε, διακριτική μεταχείριση δηλαδή λόγω της ε, εθνικής ε, ή εθνικής προέλευσης, ρατσισμός. Αυτό φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι αν αρνηθεί κάποιος να εξυπηρετήσει τους πελάτες ότι είναι φαινόμενο ρατσισμού. Μπορεί, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις όμως σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με την εσωτερική αγορά γιατί η κατοχήρωση και η προστασία των δικαιώματων είναι, ισχύει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες να χρησιμοποιήσουμε, να προσφύγουμε ε, στην ρήτρα για τα θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω ράτσας φιλετικής ε, προέλευσης ε, εθνοτικής προέλευσης. Όμως όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των πολιτών, μιλάμε για μη διακριτική μεταχείριση λόγω υπηκότητας, Αυτά άρθρο 18 της συνθήκης ε, στο κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρόλα αυτά είναι ξεκαθαρό ότι αυτό ισχύει για τα ε, νομικά πρόσωπα για κράτη. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη προσοχή πραγματεύτηκε αυτό το ζήτημα της εφαρμοσιμότητας ε, των κείμενων διατάξεων στα ε, φυσικά πρόσωπα. Για ε, κάποιους πολύ ισχυρού οργανισμούς τυποποίησης, κάποιους δημοσίους φορείς που δεσμεύονται από αυτό το δικαίωμα που πρέπει να προστατεύεται, μη διακριτικής μεταχείρισης δηλαδή, ε, λόγω της ε, γεωγραφικής τοποθεσίας. Όμως, οι μικρές, κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ε, την υποχρέωση να εξυπηρετούν όλους τους καταναλωτές, όλους τους πελάτες, το ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ενιαίας αγοράς, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και εξυπακούεται και των αγαθών. Αυτό είναι περισσότερο η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Δηλαδή, ότι είναι εφαρμοστεί αυτοί οι κανόνες ε, ε, σε σχέση με φυσικά πρόσωπα και όχι με νομικά. Το πιο καινοτόμο κομμάτι της νομοθεσίας είναι κρυμμένο μέσα στο άρθρο 20 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες. Εάν Εάν το διαβάσετε μπορείτε να βρείτε εκεί μία ιδέα σε σχέση με κάτι που μπορεί ε, που μπορεί να βοηθήσει ε, λέμε ότι δεν υπάρχουν διατάξεις διακριτικής μεταχειρίσης σε σχέση με την ε, έδρα, την γεωγραφική τοποθεσία κτλ. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για τις διαφορές όταν αντικειμενικά κριτήρια αιτιολογούν αυτή τη διαφοροποίηση. Είναι ξεκάθαρο ότι καλύπτονται οι επιχειρήσεις από αυτήν την διάταξη. Όμως, για να το πω ομά, δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα για την εφαρμογή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 8 χρόνια, δηλαδή από την ημερομηνία θέσης εφαρμογή της οδηγίας. Και ίσως υπάρχει, υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, απλώς θεωρώ ότι αυτή η διάταξη είναι απολύτως ασαφής ε, ως προς το πεδίο εφαρμογής Δηλαδή, ο στόχος ποιος είναι, να εφαρμοστεί κατά γράμμα και τίθεται το ζήτημα, μήπως είναι μάλλον προγραμματική δήλωση και όχι κανόνας που στην πράξη θα, θα ε, ε, ε, υποχρεώσει συγγνώμη, τις επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν τους πελάτες εκεί που δεν θέλουν, στις χώρες που δεν θέλουν. Εγώ θα απαντούσα, μάλλον όχι, αλλά το βλέπω από νομική σκοπιά αν θέλετε. Θα ήταν λίγο υπερβολικό ε, από πλευράς να ερμηνεύσουμε έτσι τη συνθήκη. Φυσικά κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις ε, του και σε κάποιες έκτατες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η εξαίρεση. Όμως ε, αν το δούμε ως κανόνα θα έλεγα όχι, θα απαντούσα αρνητικά. Ποιος είναι, τι σημαίνει αυτός ο κανόνας, ποιο, ουσιαστικά προωθεί τη διαφάνεια. Τουλάχιστον ο στόχος του άρθρου είναι οι επιχειρήσεις υποχρεωτικά να αποκαλύπτουν σε ποιες χώρες θέλουν να δραστηριοποιηθούν ε, και σε ποιες όχι, τουλάχιστον ε, έτσι καλύπτεται η απογοήτευση του καταναλωτή. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει την παραγγελία και μετά να του πούνε όχι δεν σα εξυπηρετούμε. Το ξέρει εξ αρχή. Δηλώνει η επιχείρηση ότι δεν επιθυμώ εγώ να, να εξυπηρετήσω πελάτε ε, στη χώρα όπου διαμένεται και πρέπει να ε, δοθεί και ε, ο λόγος για τον, της άρνησης. Για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο δεν θα αναφερθώ σε αυτά που ήθελα να πω. Ίσως ένα μόνο πράγμα. Μία επιχείρηση που κάνει πωλήσει θα, θα πρέπει να είναι στη διάθεση του δικαστικού συστήματος αν θέλει να καταθέσει μήνυση ο ε, καταναλωτής κατ' εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία του και όχι μόνο αυτό, θα, μπορεί, θα πρέπει να μπορεί να επικαλεστεί το οικείο εθνικό δίκαιο το τόπου διαμονής του ο καταναλωτής και όχι της χώρας ε, με διαφορετικό εφαρμοστό δίκαιο όπου δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο η επιχείρηση, διότι αυτό είναι ένας πιθανός φραγμός για την ενιαία αγορά. Αυτό είναι πολύ καλό για τους καταναλωτές ε, έτσι. Είναι σε μία μάλλον ασφαλή θέση οι καταναλωτές, έχουν την προστασία της χώρας προέλευσης του, κατοχυρώνεται αυτό. Κάποιες επιχειρήσεις βεβαίως το εκλαμβάνουν αυτό ως φράγμο και ίσως μεταξύ άλλων γι' αυτό διστάζουν και αποφεύγουν οι επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν σε κάποιες χώρες. Για να δούμε κάποιες προτάσεις, δράσεις σε αυτό το πλαίσιο. Carrot on the stick στα αγγλικά, ε, το καρότο ή το μαστίγιο. Ας ε, χρησιμοποιήσουμε πρώτα από όλα την πιο διπλωματική οδό να βρούμε κάποια κίνητρα ε, για να κινηθούμε ε, στα πλαίσια του τωρινού νομοθετικού πλαισίου, ώστε τα ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκαλύπτουν εξ αρχής τις χώρες από τις οποίες δεν δέχονται παραγγελίες ή ε, όπου ισχύουν πολύ διαφορετικές διαφορετικοί όροι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα στην οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Γι' αυτό το ζήτημα θα μπορούσαμε ίσως να ενισχύσουμε λίγο την νομοθεσία για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, μετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να άρει τους αντικειμενικούς λόγους για την μην χρησιμοποίηση των διατάξεων της ενίας αγοράς, ε, δηλαδή ε, πλήρη εναρμόνιση, ε, προαιρετική σύγκληση ή υποχρέωση διευθέτηση νομικών διαφορών σε άλλη χώρα. Αυτό μπορεί να, ε, ε, να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εσωτερικούς ελέγχους ε, ενδοεπιχειρησιακούς για την περιφερειακή εφαρμογή του νόμου του δικαίου ανταγωνισμού. Αυτό αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν δεσπόσα θέση στην αγορά. Υπάρχουν και αρκετές τέτοιες φυσικά. Μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να εφαρμοστεί καλύτερα διεθνώς το δίκαιο πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγόρευση Παραδείγματο χάρη ε, έκδοση αδειών με γεωγραφικούς περιορισμούς, ε, δηλαδή όσοι αδειοδότουν, όσοι χορηγούν αυτές τις άδειες λειτουργίες θα πρέπει να ε, φροντίζουν το ώστε να ισχύουν οι άδειες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι ριζική αλλαγή σε σχέση με τα όσα ισχύουν σήμερα και φυσικά εναρμόνιση των οικείων διατάξεων για τα πνευματικά δικαιώματα με το σύγκληση προς ένα ευρωπαϊκό δίκαιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στρατηγική όπου αποδίδονται οι ευθύνε, ε, blame and shame, ώστε να συμβάλλουν και οι καταναλωτέ στην καταπολέμηση ε, της διακριτικής μεταχείρισης. Ε, τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών έχουν συλλέξει ήδη τέτοιες καταγγελίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες ιστοσελίδες ε, ειδικευμένε, ε, ειδικά για αυτό το σκοπό ε, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες καταγγελίες πέρα από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προκύψουν και κάποιες ευέλτιστες πρακτικές και έτσι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και οι ενώσεις των καταναλωτών θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην πιο εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κάλλας. Πρόεδρος. Κύριε Κάλλο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κάλλας, σε σχέση με την δεσμενή διάκριση, Πάρα πολύ δύσκολο γιατί το κάνουν αυτό οι εταιρείε. Γιατί πρόκειται για τον ίδιο του τον τζίρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν. Ένα για παράδειγμα. Προσπαθούσα να αγοράσω ένα εισιτήριο για το τρένο Eurostar για να πάω από το Βέλγιο στο Λονδίνο. Δεν είχα βελγικό αριθμό, δεν μου πολλούσαν το εισιτήριο, το οποίο είναι τρελό. Όμως, ακόμη αυτό μπορεί να συμβαίνει και δεν καταλαβαίνω τι ωφελούνται από αυτό. Äh, Ευχαριστώ. Ήταν ε, πλήρης παρουσίαση. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουμε παραδείγματα τέτοια που μπορούν να συμβούν. Εγώ αγόρασα μια καφετιέρα στη Γερμανία. Η μητέρα μου ζει στη Γαλλία και ήθελε να πάρει και αυτή την ίδια καφετέρια. Ήθελα στη Γερμανία από το ίντερνετ να της την αγοράσω και έγραφε ότι δεν κάνουν παραδόσεις στη Γαλλία. Μετά μπήκα στην, ε, στο σελίδα της ε, ε, εταιρεία στη Γαλλία. Υπήρχε η καφετιέρα, αλλά στη διπλή τιμή. αγόρασα εγώ την, ε, τελικά την καφετιέρα, μια δεύτερη καφετιέρα και την έστειλα με το ταχυδρομείο στη μητέρα μου γιατί ήταν το πιο φτηνό. Είναι τέτοιες ιστορίες όλοι ξέρουμε, είναι καθημερινές, τις ζούμε και έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εταιρείε ευχαρίστως χρησιμοποιούν αυτόν τον κατακαιρματισμό της αγοράς και βεβαίως η νομοθεσία που γίνεται εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, πάντα έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε την ιστορική αγορά για τις εταιρείε. Αλλά πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια ιστορική αγορά για τους καταναλωτές. Έχουμε το άρθρο 20 της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για την οδηγία τότε και μάλιστα ε, δαπάνησα πολύ, πολύ χρόνο και πολλά νεύρα για να γίνει αυτή η οδηγία, αλλά τελικά τα καταφέραμε και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω θα μπορούσε κανείς αυτό το άρθρο 20 κατά την άποψή σας να το χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη αξία σε αυτό που μπορεί να κάνει και να φροντίσουμε ότι η ερμηνεία που θα δίνεται στην οδηγία να βελτιώνει την ε, κατανόηση των ε, καταναλωτών, να μπορεί δηλαδή να ωφεληθεί περισσότερο ο από αυτό. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή. Και μετά θα επανέλθω σε άλλε ερωτήσει, λέει ο Στα γερμανικά. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο. Δεν θέλω τώρα να σας μιλήσω για το σύνολο των παραδειγμάτων, γιατί πάρα πολλά είναι απίστευτα από αυτά που έχουμε συλλέξει, αλλά πραγματικά είναι αρκετά λογικό αυτό που γίνεται από από τις ε, πλευρά των εταιριών γιατί ουσιαστικά ο καφές είναι πολύ καλύτερο στη Γαλλία από ότι είναι στη Γερμανία. Δίνονται προφανώς μεγαλύτερη ε, σημασία σε αυτό και γι' αυτό η τιμή ήταν υψηλότερη και μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί αυτό. Ο καταγραμματισμός της αγοράς δηλαδή είναι πολύ λογικός και προφανώς αποφελείς για τις εταιρείε. Και έτσι φτάνουμε και στο πρώτο ερώτημα. Γιατί το κάνουν αυτό οι εταιρείε. Όντως πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό και επίσης το αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι. Αν αρχίσουμε από την πλευρά της επιθυμίας, θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει. Έχουμε την ιστορική αγορά, έχουμε την ψηφιακή ιστορική αγορά, και την οποία βεβαίως πρέπει να προωθήσουμε. Το πρόβλημα όμως ακριβώς είναι ότι ε, ο τρόπος που θα προχωρήσουμε μπορεί να σημαίνει ότι οι εταιρείες, και τον οποιοδήποτε λόγο, για, ακόμη και για χαζούς, ανόητους ε, λόγους, μπορεί όμως να είναι και κάτι πολύ λογικό, αλλά εν πάση περιπτώσει για τον οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να, να τις υποχρεώσουμε τις εταιρείε να κάνουν κάτι που δεν θέλουν, να, να συνάψουν δηλαδή ε, συμφωνίες ή να δραστηριοποιηθούν σε εταιρείε, σε χώρες συγγνώμη, στις οποίες δεν θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Και αυτό έχει να κάνει με σαφώ πολιτικούς λόγους. Εσείς μπορείτε αυτό να το αξιολογήσετε πολύ περισσότερο από μένα. Αλλά υπάρχουν βεβαίως και κάποια νομικά όρια και πρέπει βεβαίως να υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι. Δηλαδή και η ελευθερία της εταιρεία, η οποία βεβαίως προστατεύεται πέραν του ότι βρίσκεται και ως δικαίωμα στην συνθήκη. Ουσιαστικά λοιπόν ε, αυτό θα μπορούσε να γίνει, να υποχρώσουμε δηλαδή τις εταιρείε να υπόκεινται ε, υποχρεωτικά σε αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις. Έχουμε τώρα το άρθρο 20 το οποίο ούτως ή άλλως μιλά για το πεδίο εφαρμογής ε, Βεβαίω αυτό είναι, το αμφισβητούμενο είναι το κατά πόσο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράδοση των αντικειμένων, αλλά θα μπορούσαμε να το καταστήσουμε εφικτό και εφαρμοστέο και για την παράδοση δεδομένων, ανάλογα με τη μέθοδο που θα ακολουθήσουμε. Γιατί προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται για την, για την παράδοση προϊόντων. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια ειδική πράξη της, για την αντιμετώπιση της διακριτική διακριτικής μεταχείρισης των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Το ουσιαστικό λοιπόν πρόβλημα κρύβεται στο εξής, ότι το άρθρο 20 με την, ε, έτσι, την ε, διατύπωση που έχει, αν μπορεί να δικαιολογήσει κάποιες, ε, κάποια τέτοια παραδείγματα. Ας πούμε, σε μια τηλεφωνική συνέντευξη ρωτήσαμε μια εταιρεία γιατί ε, παρέχετε τις ε, υπηρεσίες σας μόνο στο Βέλγιο και στη Γερμανία και όχι στη Γαλλία και στις κατοχώρες ας πούμε και η απάντηση ήταν ε, στην ε, Γερμανία εντάξει μας καλύπτουν οι κανόνες και τις συνθήκες στη Γαλλία είναι αλλιώ τα πράγματα και δεν αξίζει τον κόπο είναι πολύ μεγάλος ο κόπος για να το κάνουμε αυτό να δραστηριοποιηθούμε και, και για τις κάτω το ίδιο Οπότε δεν, δεν αξίζει τον κόπο και ούτως ή άλλως έχουμε πάρα πολλή δουλειά, δεν χρειαζόμαστε άλλοι. Κάτι τέτοιο μας είπανε. Αλλά τέτοιοι λόγοι πάντα θα υπάρχουν για να μην δραστηριοποιηθεί κάποιο και να μην εξυπηρετεί μια χώρα. Ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε, α πούμε, εμεί ε, σιγά σιγά. Δεν έχουμε τι δυνατότητε ακόμα. Δεν θέλουμε να μπούμε σε άλλη αγορά ακόμα. Τέτοιες, ε, τέτοιοι λόγοι πάντα υπάρχουν. Και αυτό αναφέρεται και στη μελέτη, ότι ουσιαστικά κάθε κάθε λόγος, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, θεωρείται ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αποδεκτός από τις εταιρείε. Και αν δεν θεωρείται ε, λογικός ή εφικτός αυτός ο λόγος, θα μπορούσε η εταιρεία να βρει έναν λόγο, να, να δημιουργήσει έναν λόγο. Γι' αυτό είπα ότι το 22 της συνθήκες δεν μπορεί να επιτύχει πολλά. Ελπίζω όμως ε, πολύ περισσότερα με αυτόν τον, ότι θα πετύχουμε με αυτόν τον έμεσο ρόλο, δηλαδή ε, της παραγράφου 2 του 20 και της οδηγίας ε, για τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών. Αυτό θα μπορούσε να μπει ας πούμε σε ένα πακέτο ενημερωτικό για το ποιες χώρες μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ας πούμε, να πούμε ότι κάποιες χώρες εξυπηρετούνται, αλλά να πούμε και γιατί εξυπηρετούνται. Και θα μπορούσε κάποιος να υποχρεώσει τις εταιρείε αυτό να το γράφουν σε κάποιο πολύ εμφανές σημείο. Ε, οπότε έτσι μειώνεται ας πούμε και ο εκνευρισμός των ε, ε, καταναλωτών γιατί μέσα στα πρώτα λεπτά μπορεί να καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λάβει αυτό που θέλει να αγοράσει online. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση νομίζω ότι καλό θα ήταν να πάμε και όχι προς το υποχρεωτικό σύστημα. δεν νομίζω ότι μπορούμε να υποχρεώσουμε με κάποιο τρόπο τις εταιρείε. Ε, αυτά από μένα για τη δική σας την ερώτηση. Για την πρώτη ερώτηση τώρα, γιατί το κάνουν οι εταιρείε. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι καμιά φορά είναι χαζό. Απλώς είναι θέμα αν είναι... Ε, πώς μπορεί, αν, είναι, αν μπορεί η, Ευρωπαϊκή Ένωση να μάθει στις εταιρείε να μην είναι τόσο ανόητες αλλά το θέμα είναι η δημοσίευση των πραγμάτων. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι πιο ορατά, να είναι πιο εμφανή προς τους καταναλωτές και στα ΜΜΕ, ότι όντως υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, ότι υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι τη χάνουν διακριτικής μεταχείρισης κυρίως σε κάποια μικρότερα κρατημέλη. Αυτό δημιουργεί πραγματικά ένα πολιτικό ορόσημο και βεβαίως μπορεί να βοηθήσει να βρεθούν κάποιοι ανταγωνιστές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να γεμίσουν αυτό το κενό. Οπότε ναι, μπορούμε να πιέσουμε, ίσως αυτό είναι χρήσιμο, αλλά ίσως να μην πιέσουμε άμεσα τις εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες εκεί που δεν θέλουν να τις παρέχουν, δεν θα τις παρέχουν ε, ή και αν τις παρέχουν δεν θα είναι υψηλή ε, ποιότητας αν τις υποχρεώσουμε. Αλλά με κάποιο τρόπο να τους υποχρεώσουμε να ε, δημοσιεύσουν ότι αυτές οι εταιρείε ε, αναφέρονται και τα ονόματά του, δηλαδή, δεν παρέχουν ε, υπηρεσίες σε αυτές τις χώρες. Olga Šerleva. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εισηγή σα. Επίση, σα ευχαριστούμε και για τα όσα ενδιαφέροντα μα είπατε για την πρώτη με ερώτηση. Αλλά έχω και μια συμπληρωματική. Για αυτή την μελέτη αναφέρατε ότι ένας από τους λόγους της κατάτμισης της αγοράς είναι οι διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τους παρόγους τέτοιων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από χώρα σε χώρα. Τι έχετε να πείτε, επί τη βάση της μελέτης. Ναι, ναι, θέλω για να... και εγώ να κάνω την ε, ερώτηση. Αυτό που κάνει το Eurostar σε σχέση με κάποια εταιρεία που θέλει να μπει στην αγορά αυτό ε, αποτελεί και διακριτική μεταχείριση επί τη βάση της ε, ε της εθνικότητας, της καταγωγής, γιατί αν θέλω να ταξιδέψω από τις Βρυξέλλες στο Λονδίνο δεν μπορώ να πάω με άλλο τρόπο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι δεν μπορώ να το κάνω επειδή είμαι Εστονή υπήκος. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί οι άλλοι μπορούν και εγώ δεν μπορώ, οι Βέλγες μου μπορούν. Οπότε έχουμε ένα καινούριο νέο συρθέντα στην αγορά. Καινούργια εταιρεία. Τι θα γίνει, θα έχουμε αυστηρότερους όρους και κανόνες που θα επιβληθούν. Um, Έχετε άλλες ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Προσέξτε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι είπατε για το δικαίωμα της επιχείρησης να μην πάσχει τις σχετικές ε, υπηρεσίες σε σχέση με την προτίμηση του καταναλωτή για τις ε, διασυνοριακές. Και δεν θέλουμε να καταλήξουμε στο να αναγκάζουμε τις εταιρείε να παρέχουν τα πάντα παντού και μετά μπορεί κανένας να αγοράσει πουθενά με κανένα τρόπο μια μηχανή του καφέ. Νο θα ήθελα να αγοράσει και την πιο ακριβή. Οπότε, να. Και κάποια παραδείγματα έχουμε γιατί μπορεί να μην υπάρχουν ε, πάρα πολλέ επιλογέ για μήνυμα του καφέ, σαν το καρότο που ότι προσφέρει στην εταιρεία, ή α πούμε τι γίνεται. Γιατί από μια Εστονή δεν δέχεται η εταιρεία την πιστοτική κάρτα. Payment systems um, in Estonia, which I know has got very good e-health. Okay. Ενώ από την άλλη μεριά ανθεί το σύστημα ηλεκτρονικής ε, δημόσιας ε, στην ε, Εστονία. Να, και δεν μπορώ να πάω καν εκεί στην ε, Εστονία να πάω φάρμακα σε φαρμακείο δεν έχω αυτή την ηλεκτρονική κάρτα τη σχετική με το σύστημα υγείας. Να, που υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί φραγμοί. Αυτό ήθελα να σας πω. Οπότε θα πρέπει για να ωφεληθούν οι καταναλωτές να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες και έτσι να επικεντρωθούμε στο πώς θα ωφεληθούν και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. ιδίω με ενδιαφέρει αυτό εδώ ο κατάλογος που έχετε για τα διαφορετικά καρότα ή μπαστούνια. Να λέτε εδώ πέρα τι μπορεί να γίνει για την νομοθεσία σχέση με τα δάνεια, για το δίκαιο του ανταγωνισμού. Για πέστε μου. Τι είναι με τι απαγορεύσει σε κάποιε υπηρεσίε peer to peer όπω το Uber. Γιατί κανείς δεν μπορεί λοιπόν να σπάσει την αγορά και να μπορέσει να προσφέρει άλλου είδους υπηρεσίες σε σχέση με τις παραδοσιακές. Να κάνει αυτό και, και όχι να υπάρχουν αυτές οι απαγορεύσεις. Άλλη μια ερώτηση όσον αφορά το κοινό δίκαιο των πωλήσεων. Γιατί έχουμε όλο ένα και χειρότερες εμπειρίες των καταναλωτών Ναι, δεν θα πρέπει να τους ε, απογοητεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές. Well, thank you again for this question. Um, I start... Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, λέει ο κύριος Σουλτενόλκε. Ξεκινώ από το τέλος των Σουλτενόλκε. Είπατε για το δίκαιο των πολίσεων. Εγώ συνεργάστηκα με κάποιον από τους πιο δυσηγητές, οπότε δεν είμαι και τόσο ουδέτερος. Έκανα και αυτή τη μελέτη βιώσιμου. πάντως, μπορώ να σας πω τα εξή. Είναι καταφατική απάντηση, έχετε δίκιο, ισχύουν αυτά. Αλλά δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με κοινικό τρόπο. Οι καταναλωτέ. δεν, δεν δέχονται. Δεν εξετάζουν μάλλον το τι δικαιώματα ακριβώ έχουν. Άλλα του ενδιαφέρουν. Να δούμε βέβαια πώ θα βοηθήσουμε τι επιχειρήσει. Προστατεύοντα και τον καταναλωτή. Πάντω το δίκαιο των πολίσεων έχει τόσο ψηλό στάνταρ ώστε θα μπορούσε ο καταναλωτής να ενεργεί εμπιστευόμενος αυτή είναι ακριβώς την κοινωνική νομοθεσία άσχετα με τα όσα προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο. Και αν αυτό αποτελεί όμως φραγμό στην ενιαία αγορά και την ενιαία ψηφιακή αγορά, το, ο φραγμός είναι τα διαφορετικά ενοχικά δίκαια, τα δίκαια των συμβάσεων και τότε θα πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη με την προστασία ή θα πρέπει να έχουμε και άλλου είδους μέσα προστασίας. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι προσέγγιση νομοθεσιών, εναρμόνιση των διατάξεων. Όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες peer-to-peer και την περίπτωση της Γιούμπα, έχουμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες όπως την ελευθερία του να παρέχει κανείς υπηρεσίες που όμως έχουν κάποιους περιορισμούς και όρια που δεν είναι και λίγα. Αυτά αποτελούν νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μιλάμε εδώ για την δημόσια ασφάλεια, για προστασία του καταναλωτή και άλλες αρχές που αποτελούν περιορισμό της ελευθερίας. Δεν έχει γίνει ίσως μέχρι τώρα βαθιά ανάλυση για να το λάβει αυτό υπόψη. Γιατί τα κράτη-μέλη δικαιούνται να καθορίσουν τι θα ισχύσει όσον αφορά της, ε, ας πούμε, της υπηρεσίας μεταφοράς όπως, όπως το U-Ban. Άρα είναι εδώ εθνική αρμοδιότητα. Άπαξ και δεν έχουμε διατάξεις του κοινωτικού δικαίου όσον αφορά την μεταφορά μεταξύ Τώρα όσον αφορά τις πιστοτικές κάρτες, την κάρτα για τα φαρμακεία, να, μου θυμίζει τώρα το τι γίνεται όσον αφορά τις εξαιρέσεις των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται κατεπηγόντως, όσοι πήγονται περιστατικά. Και εδώ ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα μπορούσε σε κάποιες κατεπίγουσες περιπτώσεις να αναγκάσει τα εστονικά φαρμακεία να πωλήσουν σε κάποιον και ας μην έχει την κάρτα που είπατε. Τώρα σαν για το Eurostar. Δεν ξέρω ότι έχουμε εδώ πέρα διακριτική μεταχείριση βάσει της εθνότητας, της, της καταγωγής. Περισσότερο επί τη βάση του πού κατοικεί κανείς. Γιατί από όπου και να είστε θα πρέπει να έχετε μόνιμη διαμονή ή έστω προσωρινή διαμονή σε αυτή τη χώρα, Αν εθνικό εθνικότητας. Αν είναι θέμα εθνικότητας τότε είναι μεγάλο το πρόβλημα. Διακριτική μεταχείριση λόγω του μόνου γεγονότος ότι κάποιος προέρχεται από κάποιο κράτος μέλος, ε, αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 18 της συνθήκης και άρα είναι παράνομη άρνηση υπαρχής υπηρεσιών. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του Eurostar θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κρατικό. Εξαρτάται το ποιος κατέχει πόσες μετοχές στην εταιρεία Eurostar. Τώρα, η πρώτη, το πρώτο ερώτημα όσον αφορά τη διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ναι, ασχολήθηκε και με αυτό η μελέτη αλλά περισσότερο με κάποιες υποσημειώσεις. Και συνήθως έχουμε την ίδια ποιότητα σε διαφορετικά κρατημέλια, αλλά διαφορετικές τιμές. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πριν προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε εδώ απαρτία. Δεν θα κρατήσουν πολύ ωραία ψηφοφορίες θα αρχίσουμε στις παρατέταρτο.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 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές για τη σκληρή, πολύ σκληρή δουλειά τους και την ε, ε, πάρα πολύ καλή ε, συνεργασία που έχουμε. Θα ήθελα τώρα να αρχίσουμε την, την ψηφοφορία. Τι γλώσσα είναι αυτό. Λοιπόν, για την ασφάλεια δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκριθεί ε, η διαπραγματευτική εντολή για τον τριμερή διάλογο. Με αυτή την ψηφοφορία μπορούμε να αρχίσουμε τον τριμερή. Έχουν ξεκινήσει αυτά την προηγούμενη θητεία. Αρχίζουμε. Δεν έχουμε ψηφίσει ακόμη δύο, Όμω χρειάζονται άλλοι δύο. 29 υπέρ γιατί έλειπε μια ηλεκτρονική κάρτα. Εάν δεν έχετε την κάρτα σας, θα αντιμετρήσω την ψήφο σας, αλλά να ξέρετε ότι στα πρακτικά δεν θα καταγράφεστε, διότι είναι πλέον δημόσιες οι ψηφοφορίες και καταγράφονται τα αποτελέσματα, οπότε μην ξεχνάτε τις κάρτες σας όταν έχουμε ψηφοφορίες. Τώρα, εάν είναι πιο περίπλοκη η ψηφοφορία, είναι πολύ δύσκολο να μετρούμε κάθε φορά επιπρόσθετες ψήφους. Στη συνέχεια, αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μέλων και συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή ε, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ε, τελωνιακών και γεωργικών ρυθμίσεων. Και πάλι εξέταση και έγκριση της εντολής για την έναρξη των διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Ψηφίστε παρακαλώ. η ίδια έκφαση. 27 υπέρ 2 κατά καμία αποχή. Θα τα πούμε αργότερα εδώ στην ίδια αίθουσα στην, επιτρο... στην ακρόαση του υποψήφιου επιτρόπου. Αν είπα, όχι, λάθο, διαφορετική αίθουσα στο δεύτερο όροφο του ιδιοκτηρίου. 2Q2 στι 6.30.